Hello. Good afternoon. Καλησπέρα. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, Συνεπώ εγκρίνεται. Και στη συνέχεια έχω κάποιες ανακοινώσεις της Προέδρου. Η πρώτη έχει να κάνει με την σύνθεση της Επιτροπής Οίκων σύμφωνα με το άρθρο 209 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν γίνει κάποιε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια όσον αφορά τη νέα σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών, τη Ευρωπαϊκής και τη ΕΚΟΝ. Σύμφωνα με τι ανακοινώσει αυτέ λοιπόν σημειώστε ότι παραμένει μία κενή θέση στην Επιτροπή μα η οποία πρόκειται να καλυφθεί από τη Ρινιού, αλλά δεν έχει προτείνει ακόμα κάποιον. Και σύμφωνα με το 209 δεν υπάρχουν δικαιώματα ψήφου για μια καινή θέση και έχει προσαρμοστεί ανάλογα και το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορία. Η απόφαση για τον ορισμό των μελών στι επιτροπέ ισχύει μόνο από την ημέρα που αυτέ ανακοινώνονται στην ολομέλη από τον Πρόεδρο. Συνεπώ, δεν θα υπάρξουν τροποποίησει όσον αφορά τα μέλη τη Επιτροπή μα, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη σύνοδο στι 9 Μαρτίου του 2020. Δεύτερη ανακοίνωση για τη συνάντηση των συντονιστών την τελευταία φορά όσον αφορά τη συνάντηση δηλαδή της 22 Ιανουαρίου του 2020. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τι εκθέσει ιδία πρωτοβουλία και νοσμό εισηγητών, οι εξή ε, τίτλοι εγκρίθηκαν και έγιναν κάποιοι ορισμοί. Η πρώτη έκθεση έχει να κάνει με το σχέδιο βιώσιμη, βιώσιμων επενδύσεων στην Ευρώπη. Άρθρο 58, οι σοσιαλιστέ. Δεύτερον, ε, επιπλέον εξελίξεις όσον αφορά την Ένωση Κεφαλαγορών, πρόσβαση σε χρηματοδότηση κεφαλαίων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συμμετοχή των λιανικών επενδυτών στο ΕΛΚ. Τρίτον, αναθεώρηση του μακροοικονομικού νομοθετικού πλαισίου για καλύτερο αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία της Ευρώπης, διαφάνεια και λογοδοσία, σοσιαλιστές. Τέταρτον, ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ αποδόθηκε στο ΕΛΚΑ. Πέμπτη, ψηφιακά οικονομικά, αναδυόμενοι κίνδυνοι στα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, ρυθμιστικές και εποπτικές προκλήσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, θεσμών και αγορών. Renew. Και έκτον, εφαρμογή των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανταλλαγή όσον αφορά πληροφορίες σε φορολογικά θέματα, πρόοδος, μαθήματα που πήραμε και εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουμε ακόμα. Συνεχίζουμε τις ανακοινώσεις. Επιπλέον ορισμοί. Γνωμοδότηση για τον προπολισμό το 2021. Σοσιαλιστές. Ιδία πρωτοβουλία ε, έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης για την ε, γυραιά Ήπειρο που, γίνεται, που γυρνάει ακόμα περισσότερο. Δεν υπάρχει γνωμοδότηση. Και κάτι άλλο τώρα όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Ενισχυμένη συνεργασία με το Eurogroup. Οι συντονιστέ ενέκριναν επιστολή προ τον πρόεδρο του Eurogroup για ε, τον τρόπο συνεργασία ανάμεσα στην εικόνα και τον πρόεδρο του Eurogroup. Επίσης αποφασίστηκε να προσκαλήσουμε τον πρώτο Ευρωπαϊκό Συμβουλίου Κεντρικών Τραπεζών για μια ανταλλαγή απόψεων σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας μετά από την δημοσίευση της ετήσιας εκθεσής τους. Και όσον αφορά τη Eurostat αποφασίστηκε να προσκαλέσουμε τη Γενική Διεύθυνση της Eurostat για ένα στατιστικό διάλογο. Ε, η επιστολή πρόσκληση θα συμπεριλαμβάνει το αίτημα να υπάρξει και υποβολή μιας ε, περίληψης της πρόοδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα. Έπειτα, αποστολές της ΕΚΟΝ για το 2020, επίσκεψη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έγινε. Αποφασίστηκε και ήδη έλαβε χώρα η επίσκεψη αυτή την προηγούμενη εβδομάδα. Στη συνέχεια, αποστολή στο Βερολίνο οι συντονιστές αποφάσισαν να μην πάμε στο Βερολίνο, δεδομένου ότι μας έβαλε κάποιο περιορισμό το Προεδρείο, σύμφωνα με τις συστάσει της διάσκεψη των Προέδρων, που επιτρέπει την αποστολή, αλλά υπό τον όρο ότι δεν θα υπάρξουν συναντήσεις με την επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου. Και έτσι θεωρήσαμε ότι δεν ήταν και τόσο χρήσιμη αυτή η αποστολή και την ακυρώσαμε. Τώρα, όσον αφορά το κυλιόμενο «Don't», για να αποφασίσετε ποιοι θα πηγαίνουν στις αποστολές. Αποφασίστηκε ότι οποιαδήποτε επαναδιάθεση εδρών βάσει του συστήματος αυτού θα αποφασίζεται από τους συντονιστέ σε βάση ad hoc. Τώρα, σύγκρουση αρμοδιοτήτων. Υπήρχε το αίτημα της ΣΥΝΤΑ για δύο πρωτοβουλίε έκθεσης όσον αφορά τις εμπορικές πτυχές των μηχανισμών ε, διευθέτηση ε, διασυνοριακά του άνθρακα και αποφασίστηκε όπως πρότεινε και ο Πρόεδρος ότι η ΕΝΒΗ θα είναι η αρμόδια επί ουσίας και ΙΝΤΑ και ΕΚΟΝ θα γνωμοδοτήσουν ως δεδεμένες επιτροπές. Επίσης για το πρόγραμμα ε, πυρογνωμόνων αποφάσισαν οι συντονιστές για ένα τέτοιο πρόγραμμα κυλιόμενο ε, πυρογνωμόνων όσον αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες σε σχέση με την πράσινη οικονομία. Έπειτα για την ε, οικονομική διακυβέρνηση. Υπάρχουν δύο έγγραφα στα πλαίσια των ε, δημοσιονομικών κανόνων που ζητήθηκαν για τον Μάιο του 2020. Έλεγχος τώρα κατεξουδότηση πράξης. Έχουν εντοπιστεί τρία θέματα που είναι το MLD, το CRR και το IFRS που εγκρίθηκαν. Η προτεραιότητα θα δοθεί να οργανώσουμε κάτι μαζί με την ΛΥΜΠΕ για την ε, καταπολέμηση Τη νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τώρα, ακρόασης με ειδικού. Θέλουμε και εγκρίθηκε ακρόαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έπειτα με το ελεγκτικό συνέδριο οι συντονιστές ε, πρέπει να στείλουν τις προτάσεις τους πρώτον για θέματα που έχουν να κάνουν το πρόγραμμα εργασίας του Ελεκτικού Συνεδρίου για το 2021 δεύτερον εκθέσεις που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στην Επιτροπή μας σε μια ομάδα εργασίας μέχρι την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου παρακαλώ στη Γραμματεία. Όσον αφορά τον Brexit αποφάσισαν οι συντονιστές για γνωμοδότηση από κοινού ΑΦΕΤ Ίντα όσον αφορά την εντολή για τις μελλοντικέ σχέσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο και δόθηκε στους σοσιαλιστές. Κατευθυντήριες γραμμές τώρα όσον αφορά την ε, πρόσβαση σε τεχνικές συναντήσεις, οι τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές επιβεβαιώνονται. Και η τελευταία ανακοίνωση έχει να κάνει με μία ενημέρωση όσον αφορά τους τριμερείς διαλόγους που έχουμε. Τώρα έχουμε ένα τριμερή διάλογο που αφορά την ε, ε, τους αντισαμβελόμενους, την ανάκαμψη και την εξυγίανση των αντισυμβελόμενων. Εγκρίθηκαν διάφορα πολιτικά ζητήματα και δόθηκε εντολή σε τεχνικό επίπεδο για τα υπόλοιπα. Συζητήσαν επίσης και το δεύτερο επίπεδο όσον αφορά την ανάκαμψη των αντισυμβαλόμενων και την χρήση της αύξησης κεφαλαίου. Τα τρία θεσμικά όργανα κατάφεραν να αντιληφθούν καλύτερα ένα στη θέση του άλλου. Και το Κοινοβούλιο εξέφρασε τις έντονες ανησυχίες όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου που μπορεί να υπονομεύσει την προστασία των κονδυλίων των φορολογούμενων και τα κίνητρα προκειμένου οι αντισαβαλόμενοι να μπορούν εκ των προτέρων να αποφεύγουν τους κινδύνους και να συμμετέχουν στην ανακάμψη και την εξηγένση. Το Κοινοβούλιο επίση ζήτησε από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια ποσοτική ανάλυση για όλα αυτά τα θέματα για να αξιολογήσουμε καλύτερα το μέγεθο και τι συνέπειε του κάθε εργαλείου που διαθέτουμε για κάθε αντισυμβαλόμενο. Ο επόμενος τριμερής διάλογος θα λάβει χώρα τον Μάρτιο, στις 17 Μαρτίου. Και τώρα περνάμε στην συζήτηση της έκθεσης που έχουμε για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2020. Και θα δώσω το λόγο στην συγκίτρια, την κυρία Λαλούκ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γαλλικά, δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω οι σχέσεις που έχει το κλιματική διάσταση με την οικονομία είναι κάτι το οποίο έχουν πει και επαναλάβει οι επιστήμονες, οι οποίοι έχουν πει ότι ο τρόπο με τον οποίο αναπτυσσόμαστε, με τον τρόπο με τον οποίο προχωράει η οικονομία μα αυτό που κάνει είναι ότι θέτει σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωσή μα στη γη. Όχι τον πλανήτη, τη δικιά μα τη ζωή σε αυτό το πλανήτη. Συνεπώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να το επαναπροσανατολίσει. Δηλαδή είπε ότι πρέπει να ξαναδούμε τις οικονομικές μας πολιτικές προκειμένου αυτές να στηρίξουν την προσπάθεια που κάνουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή να διασφαλίσουμε δηλαδή την επιβίωσή μας στην Ήπειρο αυτή και στον πλανήτη και αυτό μέσα από ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ονομάζεται η Πράσινη Συμφωνία και η οποία έχει σαν στόχο ακριβώς να μας προστατεύσει όλους εμάς Ευρωπαίους και Ευρωπαίες αλλά και τον υπόλοιπο πλανήτη με μια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγή. Σε αυτό το πνεύμα λοιπόν επαπροσανατολισμού του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου εγώ πρότεινα μια έκθεση. Η έκθεση αυτή εννοείται ότι συζητήθηκε, διαπραγματευτήκαμε ευρέως. Προσπαθήσαμε να ακούσουμε όλους τους φόβους, όλες τις ανησυχίες που μπορεί να κρύβονται πίσω από μια τέτοια από ένα τέτοιο επαναπροσανατολισμό και προσπαθήσαμε να καλύψουμε τις ανησυχίες όλων. Σήμερα λοιπόν η ανησυχία αυτή ε, προχώρησε και κάνουμε μια έκθεση όχι ιδιαίτερα οικολογική ευθυγραμμιζόμαστε σε αυτά τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως, από ό,τι φαίνεται, προς το παρόν δεν υπάρχει έγκριση από όλε τι πολιτικές ομάδες. Φαίνεται ότι μια ομάδα δεν θέλει και έχει κάθε δικαίωμα βέβαια, δεν θέλει να λάβει υπόψη ε, την ανησυχία της κλιματικής αλλαγής και άλλοι δεν θέλουν να στηρίξουν την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μια άλλη ομάδα σύμφωνα με την Επιτροπή όπου συζητιέται η έκθεση, θα καταλήξω σε διαφορετική γνωμοδότηση από την ε, έκθεσή μου. Θα είμαι λοιπόν ε, πολύ σύντομη. Θέλουμε να δούμε κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που πάντα πίεζε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει, να είναι πιο φιλόδοξη, να δούμε λοιπόν κατά πόσο αυτή τη φορά έχει τη δυνατότητα να κάνει το αντίθετο, δηλαδή τελικά να προτείνει να Κάνουμε λιγότερα από αυτά που προτείνει στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λιγότερα από αυτά τα οποία ζήτησε η ίδια η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και λιγότερα μάλιστα και από όσα ζητούν οι άλλες εκθέσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που εγκρίθηκαν ε, μέχρι τώρα. Είτε πρόκειτο για σοσιαλδημοκράτη συγητή, είτε για συγητή από το ΕΛΚ. Σήμερα, λοιπόν, πριν από πέντε λεφτά μάλιστα, πήραμε κάποιες εναλλακτικές συμβιβαστικέ προτάσεις από το ECR, τη Renew και το ELK. Εννοείται ότι θα τις μελετήσουμε αυτές τις προτάσεις, αλλά ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην έχει σαν αποτέλεσμα οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιοριστούν ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε. Σκιώδης εισηγητές τώρα. Νίκο Γκιόρεφ πρώτα. Ευχαριστώ Κυρία Πρόεδρε, ο ρόρο, έχουν περάσει κάποιες εβδομάδες από τότε που ξεκινήσαμε αυτή την έκθεση. Ήταν δύσκολο και πιστεύω ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να βρούμε καλούς συμβιβασμούς. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Προσπαθήσαμε να δείξουμε ευελιξία, να συμφωνήσουμε, να λάβουμε υπόψη πολλά από τα αιτήματά σας, αλλά δυστυχώς ελάχιστο ε, συμβιβασμούς βλέπω στην τελευταία εκδοχή των συμβιβαστικών τροπολογιών. Έχω πρόβλημα και με το περιεχόμενο και με τη μεθοδολογία και θα ξεκινήσω με το περιεχόμενο. Λέτε ότι πρέπει να επαναπροσανατολίσουμε το ευρωπαϊκό εξάμενο και ότι αυτό θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αυτό που κάνετε ουσιαστικά με τις τροπολογίες σας αλλά και με την κατεύθυνση που έχετε δώσει στις συμβιβαστικές τροπολογίες είναι ότι αναδιατάσσετε και μετατοπίζετε τελείω ε, το σημείο εστίαση ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμένου. Στο μεταξύ, η δική μα δεν ήταν σαφής. Θέλουμε να διατηρηθεί ω εργαλείο αποτελεσματικού οικονομικού συντονισμού. Φυσικά και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κάποια πράγματα και να υπάρχει κάποιο επαναπροσανατολισμό, όπω λέτε κι εσεί το εγχείρημα αυτό προς μια πράσινη κατεύθυνση. Συμφωνήσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία πρέπει να ενταχθεί, να γίνεται αναφορά σε αυτήν. Αλλά η προστίκη τώρα της Πράσινης Συμφωνίας σε κάθε άρθρο αυτού του ψηφίσματος δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Θέλουμε απλούστευση, ε, κάναμε προτάσεις, ε, αλλά εσείς δεν τις δεχτήκατε δυστυχώς και θέλησατε να αλλάξετε την εστίαση. Δεύτερον, στην έκθεση αυτή προσπαθείτε να προβλέψετε πολλά ζητήματα τα οποία δεν έχουν συζητηθεί ακόμα εδώ και τα οποία είναι πολύ σημαντικά και δύσκολα. τα οποία βρίσκονται στα, στην αρχή τους αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε συζητηθεί ακόμα το κατώτατο εισόδημα, το σύστημα για την ανεργία. Ε, το να τα εντάξουμε όλα αυτά και να τα βάλουμε ως σημειοστίαση εστίασης του Ευρωπαϊκού Εξαμενού δεν μας βρίσκει σύμφωνος καθόλου. Οπότε, εν συντομία, από όψη περιεχομένου, δεν είναι χριστουγεννιάτικο δέντρο αυτό. Δεν μπορούμε να βάλουμε πάνω οτιδήποτε γνωρίζουμε ό,τι συζητείτε και ό,τι κυκλοφορεί ε, είτε η σημερινή μορφή της Πράσινης Συμφωνίας είτε άλλες ε, προτάσεις διότι για να δείξουμε ευθύνη ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διατηρήσουμε την αρχική εστίαση ότι χρειαζόμαστε σωστή χρηματοδότηση και ισορροπίες γιατί εσεί αναφέρεστε στις ανισορροπίες από την πλευρά του πλεονάσματο, αλλά ε, πρέπει να αναφέρουμε και τις ζημίες επίση και τα ελλείμματα και όλα τα σχετικά προβλήματα. Επίση τώρα για θέματα μεθοδολογικά. Εμείς ανέκαθεν είχαμε πρόβλημα σε όλες αυτές τις εβδομάδες ε, λόγω της καθυστερησμένης άφηξη των συμβιβαστικών τροπολογιών μετά από την τελευταία συνάντηση σκιωδών την Πέμπτη ε, θέλαμε μέχρι την Παρασκευή το αργότερο να έχουμε τη νέα εκδοχή των συμβιβαστικών τροπολογιών. Ενώ τις λάβαμε τελικά σήμερα στις 4 παρα 10, στις 3 ε, και 4. Ενώ ξεκινούσαμε στις 4. Ε, ο Ρορ δεν πρέπει να σας εκπλήσει που αποφασίσαμε βάσει των εμπειριών μας των τελευταίων εβδομάδων και λόγω του ότι δεν λάβαμε τις συμβαστικές τροπολογίες την Παρασκευή να συγκαλέσουμε μία συνάντηση για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια νέα εκδοχή συμβαστικών ε, τροπολογιών που σας στείλαμε πριν από λίγο. Θέλω να σας παρακαλέσω και εσάς και ε, τα κόμματα της αριστεράς. Ρίξτε μια ματιά. Θα δείτε ότι πολλές από τις αρχικές σας προτάσεις περιλαμβάνονται στις δικές μας ε, νέες εκδοχές και εξακολουθώ να ελπίζω ότι θα καταφέρετε να συμφωνήσετε για τα ζητήματα αυτά και μετά θα μπορέσουμε να κάνουμε να φτιάξουμε ένα σωστό και αποτελεσματικό ψήφισμα για το ευρωπαϊκό εξάμενο. Δεν θα είναι ε, έγκαιρο αν δεν το φτιάξουμε μέχρι το Μάρτιο. Δηλαδή η άποψή μας μπορεί να έρθει πολύ αργά αν δεν τα καταφέρουμε μέχρι το Μάρτιο όταν θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό στο Συμβούλιο. Οπότε ελπίζω να αντιμετωπίσετε το θέμα με λογική αποτελεσματικότητα και ευθύνη και με αυτή την προσέγγιση ε, ελπίζουμε να δεχτείτε τις νέες συμβαστικές μας τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ε, σκιώδης από το Ρενιό, Εγγεν Άξιο Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, ε, κυρία εισηγήτρια, Θέλω να ευχαριστήσω θερμά και την εισηγήτρια και τους βοηθούς ε, και όλους τους κοιόδους εισηγητές για την καλή συνεργασία, τουλάχιστον σε ανθρώπινο επίπεδο. Παρότι εδώ απόψη πολιτικού περιεχομένου της εκθέσεις υπάρχουν διάφορες απόψεις. Εμείς έχουμε πει καθαρά, αξιολογώντας αυτή την έκθεση, ότι για μας είναι μια αφετηρία ε, η οποία δεν είναι πολύ ισορροπημένη. Δυστυχώς η έκθεση αυτή δεν είναι έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως θα θέλαμε, αλλά προεκλογικής εκστρατείας, ε, η οποία έχει περάσει όμως. Αυτή τη στιγμή ε, κάνουμε πολιτική όλοι μαζί για την Ευρώπη. Δεν είμαστε σε φάση προεκλογική για, το, για τις ευρωεκλογές, οπότε θα ήθελα να εργαστούμε όπως πρέπει, όπως εργαζόμαστε παραδοσιακά, να δείξουμε, να εργαστούμε για τα τεχνικά θέματα και να δείξουμε στους πολίτες ότι παίρνουμε σοβαρά την εντολή μας. Εμείς ως Renew είμαστε αποφασισμένοι ε, και το λέω και το τονίζω ότι ε, εμείς το FAP και το Renew θέλουμε έχουμε υποβάλει τροπολογίες Μερικέ ε, δεν συμφωνούν απόλυτα με τη δική μου κατανόηση, με τις δικές μου πολιτικές ιδεολογίε. Ωστόσο, δεχόμαστε κάποια πράγματα εδώ πέρα, γιατί εδώ δεν είμαστε μόνο ως Renew. Προφανώς ε, υπάρχουν κάποιες ε, συμβιβαστικές τροπολογίες, τις οποίες και η δική μας ομάδα στις οποίες η δική μας ομάδα συνέβαλε με λογική. Αυτό σημαίνει βιώσιμη πολιτική και αυτή η πράσινη συμφωνία πρέπει να είναι βιώσιμη και να χρηματοδοτηθεί ακόμη και σε εποχές κρίσεων. Γιατί όταν θα προκύψει κρίση ε, απειλεί ε, τους ανθρώπους που ζουν στον πλανήτη μας και τον πλανήτη μας. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν εμείς ε, να κάνουμε ε, μια πολιτική η οποία μπορεί να οδηγεί σε κρίσεις και μετά ξαφνικά να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το σενάριο που προκύπτει. Γι' αυτό υποβάλαμε αυτές τις εναλλακτικέ ε, συμβαστικές τροπολογίες, τις έχετε λάβει και ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους από τους Πρασίνους και τους Σοσιαλιστές να διαβάσουν τις ε, τροπολογίες αυτές και να καταλάβουν ότι υπάρχει μια γραμμή όπου μπορούμε να συνεργαστούμε. Κατά την άποψή μας έτσι συμβαίνει και θα ήθελα στο μέλλον να γίνουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά, να μην ε, εργαστούμε με τον ίδιο τρόπο και ήθελα να πω τι θέλει η Επιτροπή. Ζούμε σε ένα πολιτικό σύστημα κατακρεματισμένο και καλό θα ήταν η Επιτροπή να έχει συγκεκριμένες ε, προτάσεις. Εγώ είμαι άμεσα ε, εκλεγής ερετός και πρέπει να εφαρμόζω την βούληση του λαού και των ψηφοφόρων μου και όχι της Κομισιόν. Οπότε δεν είμαστε σε προεκλογική εκστρατεία. Α εγκαταλείψουμε αυτή την ιδέα. Α πάρουμε, ας λάβουμε υπόψη μα ε, τη βούληση των πολιτών και τα επιστημονικά στοιχεία, ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε να βρούμε μια κοινή γραμμή. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Και το πρόγραμμα της Κομισιόν ψηφίστηκε από αυτό το κοινοβούλιο, ε, για να το πούμε καθαρά. Επόμενος ομιλητής, επόμενος κοιόδης, Γκούναρ Μπέκ από το ID. Δεν έχουμε σχόλια. Ευχαριστώ. Ελπίζουμε να μας φωτίσει ο Θεός και το Αγίο Πνεύμα. Ο Φίλιπ Λάμπερτς, παρακαλώ από τους πράσινους. Καλησπέρα, θα μιλήσω αγγλικά. Σε κανονικές εποχές οι εκθέσει του εξαμένου δεν αξίζουν τη μελάνη που ξοδεύεται για αυτές. Ό,τι και να πει το κοινοβούλιο, κανείς δεν ενδιαφέρεται εκτός από αυτήν εδώ την αίθουσα και είμαι σοβαρός. Ακόμη και εδώ, ε, συνάδελφοι από την Επιτροπή ΕΚΟΝ δεν ενδιαφέρονται για το τι έχουμε να πούμε εμείς για το εξάμενο. Το εξάμενο συνεχίζει την πορεία του χωρίς να λαμβάνει υπόψη την άποψη του Κοινοβουλίου. Και το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν. αν η έκθεσή μας ε, είναι ανόητη, ε, δεν υπάρχει κίνδυνος ακόμα και αν τη γράψουμε με τεχνητή νοημοσύνη και αν πειραματιστούμε, διότι ουσιαστικά ε, οι παραδοσιακέ θέσεις του Renew, του ΕΛΚ, των σοσιαλιστών, του ID, αν τις βάλουμε όλες σε έναν αλγόριθμο και γράψουμε μια έκθεση, δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτή την έκθεση, γιατί βρισκόμαστε σε μια ε, ιδιαίτερη εποχή. Έχουμε έναν επαναπροσανατολισμό των παραδοσιακών πολιτικών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε ενδεχομένω ε, θα ήταν η κατάλληλη στιγμή το Κοινοβούλιο να, επισημάνει, σημάνει τη συμφωνία, η διαφωνία του με τι νέε πολιτικέ τη Κομισιόν. Τώρα, επί τη ουσία, πρέπει να κάνουμε μια επιλογή. Είτε θα θεωρήσουμε ότι κύριε απειλέ προ την κοινωνία, προ τι κοινωνίε μα είναι ο συνδυασμό. Ε, ε, της περιβαλλοντικής ε, και της κοινωνικής ορολογιακής βόμβας και έτσι θέλουμε αυτές οι απειλές ε, να μας καθοδηγήσουν στο να χαράξουμε πολιτική ή πιστεύουμε ότι η κύρια απειλή, ο κύριος κίνδυνος για τις κοινωνίες μας είναι η δημοσιονομική απειθαρχία. Να σας πω, το καλοκαίρι του 1940 όταν ο Winston Churchill κοίταξε τις δημοσιονομικές ε, παραμέτρους ε, δεν θα είχε συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Χίτλερ διότι οικονομικά δεν είχε νόημα ούτε δημοσιονομικά αλλά υπήρχε κάτι πολύ πιο σημαντικό που διακυβευόταν και πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση. Όχι ότι έχουμε κάποια απειλή βέβαια σαν τον Χίτλερ, αλλά οι κοινωνίε μα πραγματικά βρίσκονται σε κίνδυνο και έτσι πρέπει να αποφασίσουμε τι θα καθοδηγήσει τις ε, πολιτικέ μας στο άμεσο μέλλον. Και αυτή ουσιαστικά είναι η συζήτηση. Καταλαβαίνω το ECR, το ELK, το Renew που λένε, που λένε πώς να το πω, το εξάμενο θα πρέπει να μα βοηθά να συγκλίνουμε δημοσιονομικέ και οικονομικέ πολιτικέ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτή την ιδέα. Το καταλαβαίνω και συμφωνώ. Συμφωνώ γιατί έχουμε ένα κοινό νόμισμα, μια ενιαία αγορά, χωρίς ομοσπονδιακό κράτο, οπότε χρειαζόμαστε εργαλεία πράγματι σύγκληση. Και το εξάμεινο είναι ένα τέτοιο εργαλείο. Δεν διαφωνώ λοιπόν με αυτό. Δεν πρέπει να το καταλήψουμε ως ιδέα. Ωστόσο, όπως είπε η Ορόρ, ο δεσμός μεταξύ των οικονομικών μα πολιτικών και των απειλών και ενδεχομένω των λύσεων προ αυτέ τι απειλέ είναι αρκετά σαφή. Δεν μπορεί λοιπόν να πει α κάνουμε από μια πλευρά το εξάμεινο και μετά την πράσινη συμφωνία σε άλλο επίπεδο. Αυτά τα πράγματα πρέπει να συντονιστούν. Και εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι τη συζήτηση. Πόσο ευθυγράμμιση θέλουμε. Και φυσικά υπάρχουν και διαφωνίε μεταξύ μα. Είναι σαφέ. Εγώ είμαι χριστιανό ε, και θα έπρεπε να πιστεύω σε θαύματα, αλλά δεν πιστεύω ότι γίνονται θαύματα στην πολιτική. Για μένα θα ήταν θαύμα αν το κοινοβούλιο στο νέα ισορροπία που προσπαθεί να βρει ε, αντικατόπτριζε την βούληση της Νέας Επιτροπής. Δεν μου κάνει λοιπόν καθόλου έκπλεξη ε, ο τρόπος που συζητήσαμε στη συναντήση των σκιωδών. Από όσο κατάλαβα δεν προτείνεται καμία συμβιβαστική. Φυσικά θα τα δω, δεν είμαι μέλος γραμματείας, αλλά πρέπει να δείξουμε κάποια σοβαρότητα. Είτε θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως βάση συζήτησης, είτε όχι. Και αν όχι, Ας ψηφίσουμε αύριο εδώ στην ΕΚΟΝ ε, ε, με ονομαστική ψηφοφορία. Και... Αλλά αν θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση σοβαρή, ε, χρειάζεται να του δώσουμε κάποιο χρόνο. Αυτά. Οπότε είμαι λίγο απογοητευμένο. Όχι έκπληκτο, αλλά απογοητευμένο που πράγματι φαίνεται να φυσάει νέο άνεμο από τον Περλεμόν, πολύ κοντά. Μερικέ εκατοντάδε μέτρα από εδώ. Και σε πολλέ επιτροπέ φαίνεται να φυσάει νέο αέρα, όπω και στην Έμβη. Αλλά αυτός ο άναμος, ε, όπως φαίνεται, δεν ε, παρισφρεί από τις πόρτες ε, αυτή της αίθουσα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε καλή μόνωση, βέβαια. Αλλά εγώ θα ήθελα να μπει λίγο φρέσκος αέρας, να σου πω την αλήθεια. Οπότε εγώ είμαι διατεθειμένος να συζητήσω, να δούμε αυτές τις νέες συμβιβαστικέ. Αλλά πρέπει να μας δώσετε χρόνο. Αν δεν μας δώσετε χρόνο, τι να σας πω. Οι αριθμοί είναι εκεί. Ε, εντάξει, πλειοψηφία μπορεί να βρεθεί και εδώ στην ΕΚΟΝ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ τα έχω συνηθίσει αυτά, μπορούν να συνεχιστούν για μερικά χρόνια, ακόμα μέχρι να αλλάξουν αναγκαστικά. Thank you. Now, uh, Ευχαριστώ. Ισιάρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είχαμε πολλές ενδιαφέρουσε συζητήσει τις τελευταίες εβδομάδες με τους κοιόδες συζητητέ, αλλά φοβάμαι ότι ούτε ισορροπία καταφέραμε να βρούμε, ούτε και μια καλή έκθεση. Από την αρχή ήταν σαφές ότι υπήρχαν σημαντικές διαφωνίες για το πώς η Πράσινη Συμφωνία θα αντικατοπτρίζεται στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πώ θα συντονίσουν τις οικονομικές πολιτικές και τις δημοσιονομικές τους, εγώ νομίζω ότι τα πράγματα πρέπει να παραμείνουν. Χωρίς να σημαίνει βέβαια να παραμείνουν ω έχουν, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσουμε την πράσινη συμφωνία, αλλά για μένα η κόκκινη γραμμή είναι ότι αν οι πράσινες επενδύσεις και οι πολιτικές πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο εξάμεινο, τότε υπό τους σημερινούς δημοσιονομικούς κανόνες, όπως συμβαίνει και με άλλες δημόσιες δαπάνες και με τους σωστούς δείκτες. Αλλιώς, χρειαζόμαστε νέες πράσινες επενδύσεις και νέους κανόνες. Δυσκολευόμαστε να βρούμε πόρους για τη χρηματοδότηση της Πράσινης Συμφωνίας και θα συνεχίσουμε να έχουμε δυσκολίες αν δεν εξηγιανθούν τα οικονομικά των χωρών μελών. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, τελικά αντί να ακολουθήσουν κάποιες ρεαλιστικές προσεγγίσεις, οι περισσότεροι συνάδελφοι από τη μία πλευρά βέβαια του ημικυκλίου αποφασίζουν κάτι άλλο. Όμως οι συνθήκες λένε αυτά που λένε και μιλάνε για την Ευρωζώνη. Οπότε νομίζω ότι αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Οι συνάδελφοι από το ΕΛΚ βέβαια ήταν πιο επικοδομητικοί οι επικρίσεις όσον αφορά τον φορολογικό ανταγωνισμό, την ενέργεια και άλλα τέτοια είναι εκτός πεδίου εφαρμογή. Δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση. Και άλλα πράγματα βρίσκω απαράδεκτα, το ότι αναφέρεται η ανεργία ε, με ένα μακροοικονομικό ταμείο για την ενεργεία, η ένταξη στο κοινοτικό κεκτημένο, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έντις, όλα αυτά πιστεύω ότι θα καταλήξουν σε αρνητικό αντίκτυπο και κίνητρα και δεν θα είναι υπέρ. Συνεπώς δεν συμφωνώ με την προσέγγιση της εισηγήτριας. Ε, θα καταψηφίσω τις περισσότερες από τις προτάσεις της. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Χωσέ Κουσμό. Γκουε. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. επειδή εργάστηκα για αυτή την έκθεση και επειδή ήμουν τμήμα της ομάδας που αναμφίβολα έκανε τις περισσότερες υποχωρήσεις για να φτάσουμε σε αυτές τις συμβιβαστικέ τις οποίες φτάσαμε, το οποίο είναι και κάπως φυσιολογικό, πραγματικά με λυπεί που βλέπω ότι οι ομάδες δεν είναι διαθέσιμες να κάνουν ε, συμβιβαστικές και να βρουν επικοδομητικές λύσεις. Αναγνωρίζω, για παράδειγμα, το Renew έκανε προσπάθεια τέτοια, έκανε πραγματικά ε, υποχωρήσεις σε σχέση με τις αρχικές της θέσεις και ε, ήταν και μια ομάδα η οποία επέβαλε πολλές ε, τροπολογίες σε κάποιες από αυτές τις συμβιβαστικές, κάποιες από αυτές δεν μας άρεσαν και πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι το νόημα των συμβιβαστικών. Το πρόβλημα είναι πως άλλες ομάδες ε, στην ουσία ήθελαν μέσω των συμβαστικών να ξαναγράψουν την έκθεση και αυτό είναι λίγο παρατραβηγμένο. Δεν νομίζω πως ε, είναι σωστό αυτό. Βεβαίως οι ομάδες έχουν η καθεμία το βάρος τους, αλλά δεν ε, υπάρχει έτσι κι αλλιώς απόλυτη πλειοψηφία. Εν βάση περιπτώσει, με κάποιο φόβο βλέπω και διαπιστώνω ότι Ορισμένε ομάδε, διατυπώσει τι οποίε ήδη έχει εγκρίνει το Ευρωκοινοβούλιο, όπω για παράδειγμα είχαμε στην περίπτωση του προβλήματο ε, ε, ε, του φορολογικού ανταγωνισμού και του φορολογικού dumping, πράγματα τα οποία υπόθηκαν εδώ και εγκρίθηκαν με αρκετά μεγάλε πλειοψηφίε και μετά και στο Στρασβούργο εγκρίθηκαν, δεν μπήκαν, δεν μπόρεσαν να μπουν στι συμβιβαστικέ ούτε κάνουμε τα ίδια την ίδια ακριβώ διατύπωση. δηλαδή, Σπερασπίσαμε την ιδέα ότι θα έπρεπε να υποχωρήσουμε Μάλλον, διατυπώθηκε ιδέα ότι πρέπει να υποχωρήσουμε σε σχέση με διατυπώσεις που είχαμε ήδη κάνει. Το ίδιο για τα, έγινε για τα BEPS, αλλά και για την περίπτωση του πράσινου ε, συμφώνου. Γι' αυτό λοιπόν η ομάδα μου βρίσκεται σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη κατάσταση να υποστηρίζει τις παραθέσεις ε, από παρεμβάσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εμείς δεν εγκρίναμε, προτάσεις ε, για το πράσινο σύμφωνο που εμείς απορρίψαμε και που πιστεύουμε πως είναι ανεπαρκές. Ε, και η ιδέα ότι αυτό το Green Deal είναι η, πολιτική μας, η αναπτυξιακή μας πολιτική και ότι ε, θα έπρεπε να εγκριθεί και εγκρίθηκε από όλες τις κύριες ομάδες στην Ολομέλεια. Πράγμα το οποίο όμως φαίνεται να είναι χρήσιμο για την προπαγάνδα, αλλά δεν είναι χρήσιμο για να θέσουμε σε εφαρμογή συγκεκριμένες πολιτικές με το βασικό ε, δημοσιονομικό όργανο που έχει στη διάθεσή της Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνήσαμε λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και απορρίψαμε μια ιδέα ότι το πράσινο σύμφωνο θα πρέπει να διέπει όλες τις ε, οικονομικές πολιτικές και αυτό σημαίνει πως ε, τα μέσα μας θα πρέπει να αυξηθούν μέσα σε αυτή την προοπτική. Δεν θα πει ε, να αυξηθούν. Δηλαδή το πράσινο σύμφωνο δεν θα αντικαταστήσει άλλα κριτήρια της οικονομικής πολιτικής που εντωμεταξύ όμως πρέπει να συζητηθούν όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και ε, την απόδοση που είχαν. Στην ουσία βλέπουμε λοιπόν ε, να περιοριζόμαστε στο να επαναλαμβάνουμε κάποια συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού ε, Συμβουλίου και Μάλιστα, όπως σας είπα, με αρκετά αμβλή τρόπο για να είμαστε στο πνεύμα της Συμβαστική. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν, έχετε ζητήσει κάτι the Ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ε, σημαντική έκθεση που πρέπει να βοηθήσει στο να οργανώσουμε και να δομήσουμε τη συζήτηση για την οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εάν δεν γίνει κάτι άλλο, κανένα θαύμα, αυτή η Επιτροπή δεν θα μπορέσει να εγκρίνει την έκθεση. Για την ώρα δηλαδή το Κοινοβούλιο δεν φαίνεται να μπορεί να έχει μία θέση για την ε, θέση και για την εφαρμογή του εξαμένου. Αυτό όμως ε, πιστεύω πως ε, μας αποδυναμώνει όλους. Σε μια φάση όπου είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να αναθεωρήσουμε τη λύση και την ερμηνεία του εξαμήνου και να βελτιώσουμε την ιδιοποίηση του εξαμήνου από όλου του ευρωπαϊκού φορεί, τη στιγμή που πρέπει να εντάξουμε τα περιβαλλοντικά και οικολογικά ζητήματα μέσα στην ίδια τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τηρήσουμε του ε, στόχου τη Συμφωνία του Παρισιού. Το κεντρικό σενάριο, όπως η διαγράφεται, είναι πως δεν έχει γνώμη το Ευρωκοινοβούλιο. Πρέπει να αναθεωρήσουμε, νομίζω. Κοιτούσα τις συμβιβαστικές ε, που έχουν συμφωνήσει το ΕΛΚ με το ΡΙΝΙΟΥ. Και με εξέπληξε ότι οι συμφωνίες που έφτασε τον περασμένο Ιούλιο η ομάδα των σοσιαλιστών με, τους, με το ΕΛΚ και με το, ε, ε, το ΡΙΝΙΟΥ για να μπορέσει να εκλέξει την Ούρσουλα Φαντρελάι, ενός πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ε, εδώ ε, περιττή. Δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά αναφορά στην ε, αναπτυξιακή πολιτική που, είναι χαρτοφυλάκιο ενός από τους επιτρόπους και μάλιστα σε αυτές τις συμβιβαστικέ εδώ δεν αναφέρεται πουθενά η απαραίτητη ανάπτυξη της, του κοινωνικού πυλώνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί συμφώνησαν την περασμένη θητεία. Εμένα η ομάδα μου είναι επικοδομητική και προσπαθεί να βρει συμφωνίες. Όμως ε, είναι δύσκολα αιτιολογήσιμο η ομάδα μου να δεχτεί ένα κείμενο το οποίο είναι πολύ κάτω από τις συμβαστικέ στις οποίες τάσαμε με τις ίδιες ακριβώ ομάδες με το ΕΛΚ και με το Ρενιού τον Ιούλιο και μάλιστα ε, επιπλέον έγινε και το ίδιο με την έκθεση για το Green Deal και για την οικολογική στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως έλεγε και ο συνάδελφος Γκουσμάν, διαγράφεται και η αναφορά στην ίδια την πρόεδρο ε, της Επιτροπής. Εδώ δεν υπάρχει καμιά αναφορά στις συμβιβαστικές στην Επιτροπή. και επιπλέον ε, φαίνεται πως το εξάμεινο δεν φαίνεται να είναι ο δρόμος για να απομακρυνθεί η δημοσιονομική ε, έλεγχος από τα κράτη. Μάλιστα θα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να μπορούν τα κράτη να κάνουν όποια δαπάνη θέλουν. Παρότι έχουν αυτό το δημοσιονομικό σύμφωνο. Αρνούνται να βάλουν αναθεώρηση εδώ, έλεγχο εδώ για τους δημοσιονομικούς κανόνες, για το Σύμφωνο Σταθερότητας ε, και Ανάπτυξης και για το, ε, τη, δέσμη, των, 6 και τη δέσμη των 2. Και φαίνεται δηλαδή ότι θέλει να μπορεί να κάνει το κράτος για να προωθήσει τις εταιρείε του και για να προχωρήσει σε διπόσια δαπάνη κάθε φορά που το θεωρεί σκόπιμο. Τι περισσότερη ευελιξία δηλαδή θέλετε να υπάρχει, απόλυτη ευελιξία χωρίς κανέναν έλεγχο. Θέλετε, ΕΛΚ και Εγώ νομίζω πως εν τέλει πρέπει να αναθεωρήσουμε εκ βάθρων αυτό το κείμενο. Είναι σημαντικό το Ευρωκοινοβούλιο να έχει τοποθέτηση. Θέλω να ε, εξέρω την εργασία της εισηγήτριας τις τελευταίες εβδομάδες και της ομάδας όλης, η οποία ε, πραγματικά ε, βοήθησε και με την ε, διευκόλυνση στις, στις συμβαστικές λύσεις και ευχαριστούμε την ΚΟΕ και τους πράσινους για τις προσπάθειες που έκαναν για να φτάσουμε σε συμφωνίες. Έχουμε κάποιες ώρες για να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία, αλλά η ομάδα μου, όπως είπα, δεν, μπορώ να, δεν μπορεί να δεχτεί μια συμφωνία που είναι μικρότερον μικρότερου βελονικούς από αυτήν που συμφώνησαν το ΕΛΚ και το ΡΙΝΙΟΥ για την ε, ανάληψη καθηκόντων της Επιτροπής και της Πρόεδρου της Επιτροπής. Καμία κοινωνική αναφορά, ευελιξία μόνο για τους πιο πλούσιους. Αυτό κάνετε με αυτές τις συμβιβαστικέ, αλλά όχι για αυτούς που το χρειάζονται πραγματικά. Όπως είπα, μένουν λίγες ώρες δεν ξέρω αν τελικά υπάρχει κάποια διάθεση για να φτάσουμε σε συμφωνία καλή την πίστη. Η ομάδα μου το έδειξε ε, την καλή της πίστη ε, εξετάζοντα και επαναξετάζοντα κάθε συμβιβαστική που προτάθηκε. Ελπίζω όμως πως το ΕΛΚ και το ΡΙΝΙΟΥ θα συνέλθουν γιατί δεν μπορούμε να εγκρίνουμε, όπως είπα, κάτι πολύ χαμηλότερο από τις συμβιβαστικές τις οποίες στάσαμε πριν από έξι μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Α, με συγχωρείτε, ακόμα κάποιος ζήτησε το λόγο. Η Μαργαρίδα Μάρκες. Συγγνώμη Μαργαρίδα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συνεχίσω από αυτά που είπε ο Ιωνάς για να ε, υπογραμμίσω ε, το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είναι πολύ σημαντικό να τοποθετηθεί για το εξάμεινο. Είπαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμφωνήσαμε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το εξάμεινο. Το κάναμε τη συζήτηση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται να αποσύρεται από τη συζήτηση. Αυτό σημαίνει αποδυνάμεση της θέσης μας και ε, μη πλήρη χρήση των αρμοδιοτήτων μας. Και το λέω αυτό ακριβώς γιατί η Επιτροπή των Προϋπολογισμών μόλις ε, ολοκλήρωσε και ενέκρινε την γνωμοδότησή της για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και εκεί περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση ε, κάποια σημεία που θέλω εδώ να σας παραθέσω πέρα από το ότι εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη νέα συμβιβαστική πρόταση που ζητήσαμε από την Επιτροπή, αναφερόμαστε στην σημασία των στόχων του ε, Παρισιού και επίσης για τη συμφωνία σε σχέση με τη ε, συμφωνία του Παρισιού. Ε, συμφωνία μάλλον, με συγχωρείτε, για τους στόχους της χιλιετίας και το συμφωνία του Παρισιού. Ε, δεν βλέπω λοιπόν εδώ ακριβώς πως η θέση αυτή της Επιτροπής των Προϋπολογισμών που ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία και γι' αυτό ακριβώς και φέρνω εδώ αυτή τη διατύπωση, γιατί ακριβώς πιστεύω πως το Ευρωκοινοβούλιο οφείλει να ε, τοποθετηθεί εδώ, να μην αποδυναμώσει τις ίδιες του τις αρμοδιότητες και ταυτόχρονα, όπως είπε και ο Ιώνας, δεν θέλουμε να υπονομεύσουμε το εξάμεινο ώστε να μην έχει πια ε, καμία σημασία. Έχει σημασία γιατί είναι ένας μηχανισμός που έχουμε στη διάθεσή μας για να παρακολουθούμε την εφαρμογή των δεσμεύσεων των κρατών μελών σε αυτά τα θέματα. Και γι' αυτό και νομίζω πως ε, έχει νόημα να μπορέσουμε να εγκρίνουμε μία τέτοια έκθεση και να συμπεριλάβουμε εδώ και τις νέες προκλήσεις ε, που υπάρχουν όπως αυτές που ανέφερε η Κομισιόν και όπως τις ανέφερε και ε, ε, ο κύριος Φερνάντες. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε έναν μηχανισμό παράλληλο για τα κοινωνικά θέματα και έχουμε το εξάμεινο και για αυτόν τον μηχανισμό θα πρέπει να επιμείνουμε και να εντάξουμε και αυτούς τους νέους στόχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, Ενίκο Γιώρη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να μιλήσω ουγγρικά. Βλέπουμε πως στις ε, πολλές ε, ε, έχουμε, αρκεί να διαβάσουμε τις τροπολογίες που έχουν υποβάλει τα κόμματα. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός τώρα. Δεν θα κάνουμε αγώνα εδώ ποιο έκανε τα περισσότερα. Όλοι ήμασταν έτοιμοι για συμβιβασμό. Και όλοι υποβάλαμε τροπολογίες. Διότι από αυτό το κείμενο θέλαμε να καταλήξουμε σε κάποιο ψήφισμα το οποίο να αντικατοπτρίζει ε, τις ε, συνθήκες που έχουμε στην Ευρώπη. Να συμπεριλάβουμε την ομάδα της Πράσινης Συμφωνίας, την κοινωνική ευθύνη, να δείξουμε τη σπουδαιότητα των κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά πιστεύω δεν μπορούμε να βάζουμε θέματα τα οποία δεν έχουν σχέση με όλα αυτά. Η φορολογική πολιτική. Ήδη στις συμβαστικές τροπολογίες θέλαμε να κάνουμε κάτι με αυτούς τους κανόνες που ισχύουν αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να αλλάξουν και θέλαμε να ληφθούν αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία στη φορολογική πολιτική. Ε, άλλο, κάτι, κάτι άλλο που μπήκε στο κείμενο χωρίς ε, ε εμείς να το θέλουμε. Ο χρυσός κανόνας, ε, λοιπόν, το δημοσιονομικό κομμάτι όταν ε, οι πολίτες μας, ξέρετε, ενδιαφέρονται για την οικονομία, διαβάζουν εφημερίδες, θέλουν ε, υπεύθυνη πολιτική, διαβάζουν ε, τις αξιολογήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και άλλων οργανισμών και διαβάζουν ότι ουσιαστικά βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. τι έχει να δείξει η Κομισιόν ουσιαστικά, τι, τι εξελίξεις μας περιμένουν, τι ανάπτυξη μας περιμένει. Ουσιαστικά μιλάμε για ε, μια εποχή χωρίς ιδιαίτερη ανάπτυξη, ε, με τελμάτωση, οπότε πρέπει να δείξουμε κάποια ευθύνη. Πιστεύω δεν μπορούμε ε, να παίρνουμε όλα αυτά τα οποία λέτε ως ε, γεγονότα απαραίτητα. Εγώ είμαι, υπέρ ε, του να συνεργαστούμε. Έχουμε, έχουμε δείξει κάποιο συμβαστικό πνεύμα. Έχουμε υποβάλει τροπολογίες υπό ένα πνεύμα συμβιβασμού και θέλουμε να δείξουμε ότι θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αντίξωες οικονομικές συνθήκες να ε, ε, έχει τη σωστή στάση για το ευρωπαϊκό εξάμενο ε, και γι' αυτό θέλουμε να συνεργαστούμε με, την, με τις αριστερές δυνάμεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η συγκήτρια τώρα, κυρία Λαλούκ. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπε και ο Ιχνωνάς. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρα. Για το ότι η έκθεση αυτή αντικατοπτρίζει μια πολιτική συμφωνία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να μιλήσω λίγο για τις διαπραγματεύσεις. Το ΕΛΚ μας ζήτησε να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Για να έχουμε κάτι με το οποίο να συμφωνούν όλοι. Το κάναμε. Έπειτα μας ζήτησε τα θέματα για το περιβάλλον να συμπεριληφθούν σε μία παράγραφο. Το κάναμε. Μα ζήτησε επίση το ΕΛΚ να μην αναφέρεται σε κάθε παράγραφο η Πράσινη Συμφωνία. Το κάναμε. Και θα μπορούσα έτσι να συνεχίσω για ώρε. Όσον αφορά ε, τα φορολογικά, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να υπάρχει συνένεση και το κάναμε και προσπαθήσαμε να συμφωνήσουμε και να συμπεριλάβουμε πράγματα ε, για τα οποία ψήφισε με πλειοψηφία το Κοινοβούλιο, αλλά φαίνεται ότι δεν φτάνανε αυτά. Τελικά και να κάναμε δεν ήταν ικανοποιημένα το ΕΛΚ. Τώρα για τις προθεσμίες. Και πάλι φτάνουμε με νέες προτάσεις. Εμείς θέλαμε μέχρι τελευταία στιγμή και ακόμα θέλουμε να πετύχουμε συμβιβασμό. Έχουμε νέες προτάσεις και μας ήρθαν αλλαγές τη τελευταία στιγμή από μια πολιτική ομάδα που έχει βέβαια κάθε δικαίωμα, αλλά είναι δύσκολο έτσι να συνεχίσουμε στι διαπραγματεύσει. Γιατί είναι πράγματα τα οποία αποφασίστηκαν την Πέμπτη. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με τους αρμόδιους για να κάνουμε νέες προτάσεις, να πετύχουμε συμφωνία και τελικά δεν βρήκαμε κανέναν από την άλλη μεριά της γραμμής. Ίσως να υπήρξαν ε, παρεξηγήσεις, κάποιοι να φύγανε, είναι απόλυτα φυσιολογικό, δεν λέω, δεν έχουμε πρόβλημα γι' αυτό, αλλά εμείς βρεθήκαμε ε, χωρίς δυνατότητες να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, η επιθυμία για συμβασμό υπάρχει και το ξέρετε πολύ καλά και πάντα θα την έχουμε. Θα μελετήσουμε αυτά που μας στείλατε και θα διαπραγματευτούμε μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν φοβούμαστε τις διαπραγματεύσεις και το δείξαμε εξάλλου αποδεχόμενοι όλα όσα ζητήσατε μέχρι τώρα. Κατά τα άλλα, δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα. Ο Γιώνας νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε κάτω από έναν συμβιβασμό ο οποίος μα επέτρεψε να πούμε τη γνώμη μας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Νομίζω ότι τελειώνουμε έτσι όχι βέβαια τη συνεδρίαση. Η συζήτηση αυτή ολοκληρώθηκε, αλλά έχουμε και άλλε σημαίε στην εμερήσια διάταξη. Ήταν τόσο έντονη η συζήτηση μέχρι τώρα. Λοιπόν, το επόμενο σημείο είναι ο έλεγχο των κατεξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών μέτρων. Έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων λοιπόν σχετικά με την κατεξουσιοδότηση πράξη για τον κίνδυνο αγοράς βάσει του κανονισμού για κεφαλαϊκές απαιτήσει και άλλες επικείμενες εξουσιοδότηση πράξης. Συνεπώς, Λοιπόν, όσον αφορά τον έλεγχο κατά εξουσιοδότηση πράξεων, πρόκειται για τη 44η τέτοια εποπτική συζήτηση και η εικόνα δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην ουσιαστική άσκηση των εξουσιών του, κυρίως για τις τεχνικές πράξεις. Αυτές οι ανοιχτές συζητήσεις αποτελούν πολύ βασικό στοιχείο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να ασκεί τον εποπτικό του ρόλο αποτελεσματικά. Έπειτα, στη νέα θητεία, η Επιτροπή ΕΚΟΝ θέλει να συνεχίσει τον επικοδομητικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Σήμερα λοιπόν συνεχίζουμε τις συζητήσεις για την οδηγία και τον κανονισμό για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει και επικεντρωνόμαστε στο θέμα του κατεξοδότηση πράξεων για τον κίνδυνο αγοράς που εγκρίθηκαν ήδη. Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο ε, γιατί συμπληρώνει την πράξη όσον αφορά τον κανονισμό, αλλά είναι και το πρώτο βήμα προκειμένου έχουμε και νέα μέτρα προκειμένου να καλύψουμε τις, ε, τους κινδύνους της αγοράς. Επιπλέον, έχουμε δύο τεχνικές ε, προδιαγραφές που συζητιώνται. Η μία πρόκειται για τις ρυθμιστικές τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά τις συναλλαγές σε ε, παράγωγα, χρωματοοικονομικά παράγοντα και δεύτερον για τα κριτήρια τα οποία καθορίζουν την περιθωριακή ευθύνη και τις λειτουργίες ελέγχου ε, για τις οποίες έχει ξεκινήσει ε, και διαβουλεύσεις η αρχή τραπεζών. Θα έχουμε λοιπόν την κυρία Ναταλή Μπέργκερ που είναι επικεφαλής της ΦΙΣΜΑ και τον κύριο Λάρς Όβερμπερκ για ε, θέματα κινδύνου αγοράς. Θα ακούσουμε πρώτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσείς εδώ θα έχετε από πέντε λεπτό ο καθένας. Πρώτα θα ακούσουμε λοιπόν για την νέα κατοξιδότηση πράξη όσον αφορά τους κινδύνους αγοράς. Και μετά θα έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις. Λοιπόν, πρώτα η κυρία Μπερζέ. Πού είναι? Εκεί. Okay. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω υπενθυμίζοντας πρώτα απ' όλα ότι η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία έχει θέσει το πλαίσιο όσον αφορά τους κινδύνους αγοράς ήδη από το 2016. Και αυτή ακριβώς είναι και η βασική αναθεώρηση που έγινε για τα χαρτοφυλάκια. Αυτό αμέσω μετά την κρίση. Μέρος της αναθεώρησης αυτής είναι δημοσίευση από την Επιτροπή της Βασιλείας κάποιων τυποποιημένων στοιχείων όσον αφορά τους κινδύνους της αγοράς. Και εμείς θέλουμε να εισάγουμε στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο προδιαγραφές τεχνικές για να καλύψουμε το πακέτο του 2016 με τροποποίησεις όσον αφορά τον κανονισμό κεφαλαικών απαιτήσεων. Όμως, οι διαπραγματεύσεις όσον αφορά τον κανονισμό κεφαλαικών απαιτήσεων είχαν ήδη προχωρήσει πολύ και ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2019 όταν ακριβώς η Επιτροπή της Βασιλείας ε, προχώρησε σε ουσιαστικές αλλαγές των προδιαγραφών. Και ο νομοθέτης αποφάσισε τότε να χρησιμοποιήσει τη νέα ε, προσέγγιση προδιαγραφών, η εναλλακτική προσέγγιση δηλαδή, προκειμένου να υπολογίσει τις κεφαλικές απαιτήσεις όσον αφορά τους κινδύνους της αγοράς για λόγους παρουσίασης στοιχείων μόνο και έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει διορθώσεις στον κανονισμό κεφαλικών απαιτήσεων που είναι αναγκαίες για να προσαρμόσουμε τους κανόνες της Βασιλείας σε ένα επίπεδο νομοθεσίας 2 τροποποιώντας ακριβώς τις προδιαγραφές για τον κανονισμό κεφαλικών απαιτήσεων. Και οι τροπολογίες αυτές αποτελούν και την ουσία της κατεξοδότησης πράξης που παρουσιάζω σήμερα. Ο λόγος δηλαδή για τον οποίο κάναμε ουσιαστικά τα στοιχεία εκείνα που δεν είχαμε κάνει αρχικά ήταν γιατί οι νομοθέτες αποφάσισαν τελικά για το πακέτο κεφαλικών απαιτήσεων όσο η διαδικασία στην Βασιλεία ήταν ανεξελίξη. Συνεπώς τώρα με την κατουξιδότηση αυτή πράξη εμείς ζητάμε για λόγους παρουσίαση στοιχείων και για λόγους εφαρμογής της βασικής αναθεώρησης του χαρτοφυλακίου για λόγους κανονισμού κεφαλαικών απαιτήσεων στα πλαίσια της νέας νομοθετικής πρότασης η οποία θα εγκριθεί αργότερα φέτος. Συνεπώς, αυτή την κατεξοδιώτηση πράξη, όλα τα θεσμικά όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν trading book θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτήν την εκτελεστική, αυτή συγγνώμη, την κατεξοδότηση πράξη για λόγους αναφοράς εκτός αν εξαιρούνται. Και ο νομοθέτης συμφώνησε για κάποια όρια όσον αφορά τις εξαιρέσεις που είναι πολύ ψηλά. κάτω από 500 εκατομμύρια σε αξία της αγοράς. Έτσι ώστε μόνο οι τράπεζες που, είναι, που έχουν ένα μεγάλο ή ένα μεσαίο χαρτοφυλάκιο συναλλαγό να προχωρούν στη διαδικασία αυτή. Υπάρχει Επίσης και η Διοργανική Συμφωνία της 13 η Απριλίου του 2016 για καλύτερη νομοθέτηση και συμβουλευτήκαμε και ειδικού για τις κατεξουδότηση πράξη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί τη διευκαιρία. Οργανώσαμε δύο συναντήσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων μας στις 13 Ιουνίου η πρώτη και η δεύτερη στις 26 Νοεμβρίου με την συμμετοχή και της Γραμματείας της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Επίσης, προχωρήσαμε και σε μια διαβούλευση με το κοινό. Είχαμε άτυπες διαβουλεύσεις, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ήθελαν να, να μας παρουσιάσουν τις απόψεις τους όταν ετοιμάζαμε την κατοξιδότηση πράξη. Πήραμε 8 απαντήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανώσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επειδή είναι τεχνικής φύσεως η πράξη αυτή, δεν θα σας εκπλήξει ε, το γεγονός ότι δεν πήραμε απαντήσεις από το ευρύ κοινό, ας το πω έτσι. Κάποιοι απάντησαν με πολύ χρήσιμες προτάσεις. Κάποιοι μάλιστα προσέφεραν και κάποιες προσαρμογές ή διορθώσεις. Κάποιοι πρότειναν καλύτερη ευθυγράμμιση του σχεδίου κατεξοδότηση πράξης με τις προδιαγραφές της Βασιλείας. Εμείς λάβαμε υπόψη μας τα σχόλιά τους στο βαθμό όπου τα σχόλια αυτά, οι προτάσεις αυτές καλύπτονται από την εντολή μας και επιμένω πάνω σε αυτό. Διότι ε, πήραμε και κάποια σχόλια που μας ζητούσαν παραπάνω προσαρμογές στην κατεξοδότηση πράξη που δεν μπορούσαμε όμως να υλοποιήσουμε εμείς γιατί δεν μας καλύπτει η εντολή που έχουμε από τον νομοθέτη. Οπότε αυτά τα σχόλια δεν τα λάβαμε υπόψη μας. Επιπλέον, εποφεληθήκαμε και από σχόλια της ε, ομάδας για τους κινδύνους αγοράς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Επί της ουσίας τώρα, οι αλλαγές που επιφέρει η κατεξοδότηση πράξη στι κεφαλαϊκέ απαιτήσει λαμβάνει υπόψη την ευαισθησία της ε, νέα αυτής εναλλακτική προσέγγισης. Και γι' αυτό φροντίζει για τους κινδύνους ε, ισοτιμιών, για τις επιχειρήσεις, ε, για τους δείκτες και για τις διάφορες επιλογές. Επίσης, προσφέρει και στάθμιση που προσφέρεται σε γενικούς κινδύνους ισοτιμιών αλλά και έκθεση σε επιστοτικούς κινδύνους. Όλες αυτές οι αλλαγές ήταν αναγκαίες για να καταλήξουμε στις τελικές προδιαγραφές που ενέκρινε και η Επιτροπή της Βασιλείας το 2019 και όπως αποφασίστηκε στις πολιτικές συμφωνίες για τις κεφαλικές απαιτήσει 2, η κατεξοδότηση πράξη λαμβάνει υπόψη τις προδιαγραφές των προδιαγραφών της ε, βασιλείας κάθε φορά που πρόκειται για αναφορές, για παρουσίαση στοιχείων. Όπως γνωρίζετε και το είπα και στην αρχή, η νομοθετική μας πρόταση για τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις 3 θα προσπαθήσει να συμπεριλάβει και τις νέες προδιαγραφές της Βασιλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δει πώς θα μπορούσαν και οι απαιτήσει για παρουσίαση στοιχείων να συμπεριληφθούν στη, στον κανονισμό και τις κεφαλαϊκές απαιτήσει. Εννοείται ότι παρατηρούμε και παρακολουθούμε και τις εξελίξεις σε άλλες δικαιοδοσίες όσον αφορά τις προδιαγραφές για κεφαλαϊκές απαιτήσει. Είχαμε κάποιες επίσης συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και που προσπάθησε να μας βοηθήσει ανταποκρινόμενη στις, ε, στη διαβούλευση που εμείς είχαμε ξεκινήσει. Θα λάβουμε υπόψη μας ε, λοιπόν τα σχόλια της Ευρωπαϊκής ε, Αρχής Τραπεζών και όλα τα άλλα που πήραμε στην νέα μας πρόταση. Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση στις αρχές αυτής της χρονιάς και πήραμε πάνω από 100 απαντήσεις. Τέλος, να ξέρετε ότι οι θεσμοί θα μπορούν να φέρουν σε πέρα τις υποχρεώσεις τους παρουσίαση στοιχείων βάσει αυτής της κατεξουδότηση πράξης, εφόσον η αρχή τραπεζών θα έχει καταλήξει σε τεχνικές προδιαγραφές με συγκεκριμένο πίνακα και οδηγίες για τη συμπλήρωση των ε, τεχνικών προδιαγραφών. Μέχρι τις 3 Ιουνίου φέτος. Οι πράξεις αυτές πάντως θα παρουσιαστούν συγχρόνως και θα υπάρξει περίοδος 6 μηνών για την εφαρμογή. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω τις δικές σας παρατηρήσεις και τα σχόλια. Ευχαριστούμε με το λόγο τώρα Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση σήμερα. Χαίρομαι που δίνει τέτοια έμφαση στις κατεξοδότηση πράξεις στο Κοινοβούλιο. Είναι τεχνικό θέμα και αρκετά σημαντικό για την υλοποίηση των ζητημάτων αυτών που αντιμετωπίζουν οι επόπτε και οι τράπεζε, Οπότε είναι πολύ καλό αυτό το έγγραφο. Δίνει μια γενική εικόνα των δύο ζητημάτων που σχετίζονται με την κατεξοδότηση πράξη, ή ε, τυποποιμένη αυτή τη προσέγγιση, η τυποποιημένη αυτή προσέγγιση, η ΣΑΚΑ και το RTS ε, για όσου διατρέχουν κινδύνους που βρίσκεται υπό διαβούλευση για τους διαχειριστές όπως είπε και η Νάταλη είχαμε και εμείς εντατικές συζητήσεις όπως είπε και η Νάταλη Όσον αφορά τα στάνταρ αυτά, τα ΣΑΚΑ, είχαμε ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα, αλλά είχαμε, καταφέραμε να το υποβάλουμε μέχρι τα τέλη του έτους ε, στην Κομισιόν. Παραμείναμε πιστοί στην αρχική πρόταση που προέκυψε την αρχική μας διαβούλευση με, με ρεαλιστικές λύσεις και πρακτικές λύσεις ε, για την αντιμετώπιση των ε, προβλημάτων ε, σε τέτοιες συναλλαγές και είδαμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και τα ζητήματα των αρνητικών επιτοκίων που αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζονται βάσει των προϋποθέσεων και τις κεφαλαίκες απαιτήσει υπό την προσέγγιση ΣΑΚΑ. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ευθυγραμμιζόμαστε με τα πρότυπα της Βασιλείας που ήταν ήδη ρεαλιστικά ως προς τις λύσεις που προσέφεραν ειδικότερα όσον αφορά τα αρνητικά επιτόκια επιπλέον δώσαμε αρκετή έμφαση σε καθορισμό προτεραιοτήτων. Αυτό είναι το πρώτο βήμα στο συνολικό μας ε, οδικό χάρτη που το δεύτερο κομμάτι για το RTS και για αυτούς που αναλαμβάνουν κινδύνους βρίσκεται ακόμα σε πρώιμη φάση διαβουλεύσεων. Οι διαβουλεύσεις θα κλείσουν την Τετάρτη. Η επικαιροποίηση στο υπαρχόντος RTS με αλλαγές στο άρθρο 72 στο CR5 χρειάστηκε να ε, φτιάξουμε ένα νέο προσέδιο όπως μας ζητήθηκε. Κάποια από τα κριτήρια που υπήρχαν ήδη στο RTS έχουν τώρα συμπεριληφθεί απευθεία στην οδηγία. Χρειάστηκε λοιπόν να επικαιροποιήσουμε το αρχικό σχέδιο RTS. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε ότι δεδομένου ότι τώρα περνάμε από τον καθορισμό των τεχνικών προτύπων στην υλοποίηση μέχρι το 2020 από τις αρχές, μεταφορά δηλαδή διεθνούς δικαίου. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι Υπάρχουν διασυνδέσεις και με το Φαραφέρντι και υπάρχουν κάποιες αλλαγές που μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιες συνέχειες μεταξύ των δύο πλαισίων που προσπαθούμε εμείς να λάβουμε υπόψη ε, στις εργασίες μας. Όσον αφορά το περιεχόμενο, η εντολή είναι αρκετά απλή ε, για να παρέχεται ένα νέο σύνολο ορισμών που σχετίζονται με πράγματα όπως η ευθύνη των ε, managers ε, και οι μονάδες εξέθεσης κινδύνου και πώς ε, αυτό επηρεάζει τους οργανισμούς μας. Επιπλέον προσπαθούμε να διατηρήσουμε την αρχική προσέγγιση που τέθηκε σε ισχύ το 2014. Προσπαθούμε να επικαιροποιήσουμε και διάφορα ελάσσονα ζητήματα. Για παράδειγμα στους κινδύνους IT που είναι όλο και μεγαλύτεροι η επικεφαλής ε, πληροφορικής και ασφάλειας πληροφορικής ε, επίσης θα πρέπει να ορίζονται ως προσωπικό να είναι συγκεκριμένοι μαζί με τον επικεφαλής του outsourcing. Το τελευταίο κομμάτι όλου αυτού σχετίζεται με τις απαιτήσει ε, αμοιβών που καλύπτεται εδώ και αφορά όλους τους οργανισμούς ανεξαρτητός μεγέθους. Έχουμε λάβει σημαντικά ε, πολλά αιτήματα από μικρούς οργανισμούς που προτιμούν ε, μια πιο απλή διαδικασία ταυτοποίησης. Αυτό αποτελεί και το αντικείμενο του εγγράφου διαβούλευσης που αφορά ε, την εφαρμογή της αναλογικότητας σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να έχουμε μετριασμένες προσδοκίες. Είναι αδύνατο να πληρωθούν όλες οι απαιτήσει. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε κοινά στοιχεία και αυτό θα ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα έχουμε τον κατάλογο αγορητών για τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Ξεκινάμε την Τανούτα Χούπνερ από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω εκ μέρους του Ατμαρ Κάρας ουσιαστικά που είναι και εισηγητής για το CRD4 και το CRR και για το CRD5 και για το CRD2 ήταν. Δεν μπορούσε να είναι εδώ. Μου ζήτησε να σχολιάσω για τρία ζητήματα και να κάνουμε έξι ερωτήσεις. Υπογραμμίζω ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί αυτή η αναθεώρηση. Τώρα υπάρχει υποχρέωση τέτοια και η δυνατότητα μιας μικρής περίοδου ελέγχου λίγων ε, μηνών δεδομένου ότι το κείμενο που υιοθετήθηκε από την Κομισιόν είναι αυτό που παρήχε η ΕΣΑΣ. Ο κύριος Κάρας θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει τους εκπροσώπους της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών που βρίσκονται εδώ μαζί μας. Χάρη σε αυτούς μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τον έλεγχο των μέτρων επίπεδου 2. Θα ήθελε επίσης να πει ότι διακρίνει πρόοδο αλλά και καθυστερήσεις και εκκρεμή ζητήματα μετά από την τελευταία με τον τελευταίο έλεγχο του Ιούνιου του 2018. Τα ζητήματα αυτά αφορούν την καταξιδότηση πράξη για τους κινδύνους αγοράς. Πιστεύει ότι αυτή η καταξιδότηση πράξη είναι συνήθιστη. Δεν συμπληρώνει, ε, ξαναγράφει ε, το CRR. Ουσιαστικά ε, στη διαδικασία επίπεδου 1 δεν είναι παρά το βήμα 1 γιατί θα, θα εφαρμοστεί ούτως ή άλλως η κεφαλαϊκή απέτηση και οι δύο ερωτήσει είναι οι εξή πρώτα απ' όλα δεδομένου ότι τα άρθρα 325 ΑΙ δεν καλύπτονταν από την εξουσιοδότηση. Η ερώτηση είναι η Κομισιόν πιστεύει ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα ότι Πώς θα γίνονται με τις νέες ε, τιμές συσχετισμού μέσω αυτής της κατεξοδοτής πράξης και και κατά πόσο αυτό θα είναι απαραίτητο και προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για ποιους λόγους η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών προβλέπει ε, ημερομηνία εφαρμογή για την απέτηση ε, αναφορά ε, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο στι 31 Μαρτίου του 2021 αντί για όχι αργότερα από τον Δεκέμβριο του 2020 όπως προβλέπεται τώρα στην κατεξοδότηση πράξη. Το δεύτερο ζήτημα σχετίζεται με το τελικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζών για τις συναλλαγές και η πρώτη ερώτηση προς την Κομισιόν είναι θα πραγματοποιήσει η Κομισιόν διαβούλευση πριν από την υιοθέτηση τη κατεξοδότηση πράξη. Είναι τη άποψη ότι οι διαβουλεύσει τη Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ήταν αρκετέ. Και η δεύτερη ερώτηση εδώ είναι η Επιτροπή μπορεί να μα αναλύσει σε ποιο βαθμό και σε ποιου τομεί θα παρεκκλίνει από το τελικό σχέδιο RTS ε, της Ευρωπαϊκής Αρχή Τραπεζών και το τελευταίο ζήτημα όσον αφορά το σχέδιο αυτό για την διαχειριστική ευθύνη και τις ε, λειτουργίες ελέγχου. Η πρώτη ερώτηση είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα μπορούσε να μας αναλύσει που το κάνατε νομίζω, αλλά ε, υποχρεώμαι να το διαβάσω, κατά πόσο θα εξετάσετε το ενδεχόμενο της αναλογικότητας να ληφθεί υπόψη ώστε να αποφευχθεί φόρτος για μικρούς, μη περίπλοκους οργανισμούς και η τελευταία ερώτηση η Κομισιόν έχει επιβεβαιώσει το αίτημα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών να παρατείνει το χρονοδιάγραμμα υποβολής μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε, πιστεύω, να μαζέψουμε όλες τις ερωτήσεις μαζί. Κύριε Φερνάντες, από τους Σοσιαλιστές. Sí, muchas gracias, Presidenta. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα απομακρυνθώ πολύ από τις ερωτήσεις κάραση της κυρίας Ντανούτα. Αντικαθιστώ και εγώ τον εισηγητή. Για τα θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτή η κατεξοδότηση πράξη για τον κίνδυνο αγοράς βάσει του άρθρου 461α θα μπορούσε να επεκτείνει τις αρμοδιότητες στο επίπεδο 2 και θα μπορούσε να επηρεάζει απευθείας τις δυνατότητες ε, συνομοθέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσφέροντας αλλαγές στο επίπεδο 1. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω κι εγώ ό,τι ρώτησε και η Ντανούτα ή ο Κάρας. Και να ρωτήσω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς τα βλέπει. Τα βλέπει όπως και εμείς, ότι δηλαδή ξεπερνάει τις αρμοδιότητές της. Και αν πιστεύει πως όχι, να μας το εξηγήσει αυτό. Επίσης, στα πλαίσια της αναθεώρησης του συνόλου των κεφαλαικών απαιτήσεων που ε, Ετοιμάζουμε τώρα, λαμβάνοντα υπόψη τι συστάσει τη Βασιλεία και περιμένοντα την νομοθετική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του επόμενου μήνε, θα ήθελα όμω στο μεταξύ να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ αναλύει εκείνη τον αντίκτυπο αυτών των κατεξουδιώτηση πράξεων για τις κεφαλαικές απαιτήσει και πώς θα επηρεάσουν αυτές το έργο μας τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μπέλη Γκάλα, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω εξ αρχής ότι καλά είναι και είναι ε, για αυτό το θέμα και μου ζήτησε, επειδή δεν μπορούσε να είναι παρούσα, να διαβάσω το σχόλιά της. Ε, το αναθεωρημένο πλαίσιο της βασικής ε, έκθεσης δημοσιεύθηκε το Ιανουάριο του 2019, αλλά δεν ήταν πολύ αργά για να εσωματωθεί στη συμφωνία του Μαΐου του περασμένου χρόνου το θέμα του κινδύνου της αγοράς είναι σημαντικό γιατί αντικαθιστά το ισχύον κείμενο επίπεδου 1. Στη διάρκεια της, της χρηματοπιστωτικής κρίσης το δημοσιονομικό πλαίσιο δεν ήταν σαφές και οι τράπεζες μπορούσαν να επιλέξουν ανάμεσα στο banking book και το trading book, ανάλογα ποιο είχε το πιο ευνοϊκό αντίκτυπο. Για να του 19 συμπεριλαμβάνει κάποιες ε, αναθεωρήσεις της εναλλακτική τυποποιημένης προσέγγισης, θεωρώ πως είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τον κίνδυνο της αγοράς. Δεν εισάγει ακόμα κεφαλαίκες απαιτήσει, αλλά οι αναφορές περί, περί των ε, κεφαλαϊκών απαιτήσεων είναι πιο ε, εφικτές και θα παρουσιαστούν τον Ιούνιο του 2020 το αργότερο. Θα ήθελα να, ξε... να θίξω την εξή ερώτηση. Η κατεξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής αναφέρει ρητά ότι δεν είναι σε θέση να καλύψει την εισαγωγή νέων ε, αξιών συνεχισμού, συσχετισμού όσον αφορά τους παράγοντες πιστοτικού κινδύνου. Ποιος, πώς θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος τρόπος να περιμένουμε την αναθεώρηση CRD-CRR για, να για να εφαρμόσουμε τη Βα... Βασιλεία 3 ή το CRR 5. Υπάρχει κάποια άλλη ε, ε, καλύτερη λύση. Για τις δύο άλλες ε, ε, RTS, για τις συναλλαγές σε παράγωγα και τον κίνδυνο για την ευθύνη των διαχειριστικών στελεχών, θα θέλαμε να δούμε τα πορίσματα πριν να αποφασίσουμε πάνω σε αυτές. Ωραία, σας ευχαριστώ. Έχουμε κάποιους ακόμα Χουάν, ε, ο, ο Γιώνας Φερνάντες θα μπορούσε να πάρει το λόγο. Όχι, δεν θέλει να πάρει το λόγο. Θα μείνουμε λοιπόν σε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ε, η Κομισιόν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ θα ξεκινήσω με το γενικό θέμα όσον αφορά το θέμα της ε, της ε, χειραφέτησης ή της ενίσχυσης, αυτή είναι κάπως ασυνήθιστη ως ε, κατεξοδότηση πράξη. Ο νομοθέτης αποφάσισε να ζητήσει από την Κομισιόν να προχωρήσει σε τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων της βασικής πράξης. Οι συνομοθέτες αποφάσισαν να δώσουν και προθεσμία στην Κομισιόν για να ολοκληρώσει αυτό το έργο και η προθεσμία ήταν η υιοθέτηση της κατεξουσιοδότησης συμπράξης πριν το πέρας του 2019. Οπότε, Κάνοντας το αυτό και υιοθετώντα την κατεξουσιοδότηση πράξη, δεν νομίζω πως ε, ξεπερνάμε τις αρμοδιότητές μας ε, ε, ή τις δυνατότητές μας. Αντίθετα, ότι τηρούμε την εντολή που μας δόθηκε από τους συνομοθέτες. Και μπορεί κανείς να δει τη συνέπεια το περιορισμό αυτό, αυτής της εντολής λόγω των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν όσον αφορά τους συσχετισμούς ε, και για την ε, θέσπιση των νέων αξιών συσχετισμού. Γιατί ακριβώς αυτό ήταν ένα ζήτημα στο άρθρο 3.2.5 EI. Ε, το εξετάσαμε λοιπόν αυτό, γιατί θα ήταν πολύ θετικό να ήμασταν σε θέση πράγματι να ορίσουμε αυτά ε, τις δυνατότητες και τις αξίες σχετισμού. Όταν όμως το κάναμε, αν και μπορούσαμε να το κάνουμε από τεχνικής άποψης, προσέξαμε να μην ξεπεράσουμε την εντολή μας και γι' αυτό ακριβώς σε αυτήν την κατεξοδότηση πράξη βλέπετε ότι δεν υπάρχει τίποτα για τις αξίες συσχετισμού. Τώρα, εφόσον η Κομισιόν δεν είχε λοιπόν εντολή να δράσει, πώς θα προχωρούσε στην πράξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του κανονισμού κεφαλαικών απαιτήσεων 3, όπου έχουμε όντως να κάνουμε μονομοθετική πρόταση και εντωμεταξύ για τις ε, συγκεκριμένους στόχους ε, των αξιών ε, συσχετισμού, θεωρούμε πως οι τράπεζες θα μπορέσουν να προχωρήσουν επί τη βάση εποπτικών αποφάσεων ή εγκρίσεων. Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο θα καθοριστεί ανά περίπτωση σε συνεργασία με τους εθνικούς επόπτες. Αλλά δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε γιατί αν το είχαμε κάνει αυτό θα είχαμε ξεπεράσει την εντολή μας και το συγκεκριμένο αίτημα των συνομοθετών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, sorry, there was a question Αχ, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Υπήρχε και μια άλλη ερώτηση που αφορούσε την ανάλυση του αντικτύπου ε, το ε, βασιλεία στις, στις απαιτήσει. Δεν μπορέσαμε να συνοδεύσουμε την ε, πράξη, την κατεξοδότηση με ε, ε, εκτίμηση αντικτύπου, γιατί δεν θα ήμασταν σε θέση να τηρήσουμε την προθεσμία που μας είχε επιβάλει ο νομοθέτης. Χρειαζόμασταν τεχνική συμβουλή και δεν μπορούσε αυτό να γίνει μέσα στο ένα πλαίσιο εξαμήνου. Είμαστε λοιπόν στην πορεία της αξιολόγησης ε, του αντικτύπου και του αντικτύπου για την ε, βασική αναθεώρηση του Trading Book για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε την νομοθετική μας πρόταση στο πλαίσιο του ε, κανονισμού κεφαλαικών απαιτήσεων επαριθμών 3. Εκεί θα βρούμε όλες τις απαντήσεις και τις αναλύσεις και μετά στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε πώς ε, και ποιες πολιτικές επιλογές θα προτείνουμε στους συνομοθέτες ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν. Αυτά όλα θα γίνουν επί τη βάση μιας πλήρους ανάλυσης αντικτύπου που φυσικά βασίζεται στη τεχνική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής που με τη σειρά της συνοδεύεται από ε, μελέτη αντικτύπου και προχωρούμε και όλα σε τη βάση των απαντήσεων που λάβαμε στο πλαίσιο της εκτεταμένης δημόσιας διαβούλευσης. Μελέτη αντικτύπου λοιπόν είναι υπό εξέλιξη και θα ετοιμαστεί, θα συνοδέψει την νομοθετική πρόταση για το ε, κανονισμό κεφαλαικών απαιτήσεων παριθμών 3. Σας ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Ναι, νομίζω πως ε, δύο ερωτήσεις ε, απευθύνονταν σε μένα. Μία αφορούσε τα δεδομένα εφαρμογής και τις απαιτήσει αναφορών, τα οποία περιμένουμε από το Μάρτιο του 2021 αντί για Σεπτέμβριο 2020. Κατά βάση πρόκειται για μια ρελεστική επιλογή, όπου με την έγκριση και την υποβολή του της κατάστασης κινδύνου του RTS θα περιμένουμε ε, ένα διάστημα τρίμηνο αλλά ε, ο κλάδος δεν μπορεί να προετοιμαστεί για μια τελική κατεξοδότηση πράξη. Γι' αυτό και δώσαμε ακόμα έξι μήνες ώστε να προετοιμαστεί η εφαρμογή, πράγμα που είναι συντομότερο από αυτό που κάνουμε συνήθως μέσα στον κύκλο αναφορών, όπου συνήθως στοχεύουμε σε 12 προετοιμασία, ώστε να μπορέσει ο κλάδος να εφαρμόσει νέες σημαντικές απαιτήσεις. Προσπαθούμε λοιπόν να κινηθούμε όσο γίνεται ε, πιο γρήγορα όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό, αλλά πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλο χρόνο για να προετοιμαστεί ο κλάδος ε, καταλήλω. Όσον αφορά τις απαιτήσεις αναλογικότητας, νομίζω πως ε, το ανέφερα αυτό στην εισήγησή μου, στο RDS όσον αφορά την ανάληψη κινδύνων ε, θέλουμε να εξετάσουμε πώς θα εντάξουμε τις πιθανές αλλαγές και την πιθανή αναλογικότητα για τις μικρότερες τράπεζες. Ένας τρόπος θα ήταν να θεσπίσουμε, για παράδειγμα, ένα πιο περιορισμένο υποσύνολο κριτηρίων που θα ισχύει για τους μικρότερους ε, παίχτες. Ε, αυτό θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος να προχωρήσουμε, αλλά πάντως δεν μπορεί να μην υπάρχουν απαιτήσει. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει γιατί το πρώτο επίπεδο πρέπει να αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω κανέναν άλλο να ζητά το λόγο, να θέλει να υποβάλει ερωτήσεις, οπότε ε, τώρα πιστεύω πως κλείσαμε και την σημερινή μας συνεδρίαση και θα συνεδριάσουμε και πάλι αύριο στις 11 το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ.